Uh, good afternoon, colleagues, and welcome back to our committee. Um... Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και πάλι. Χαίρομαι πολύ που σήμερα για την απογευματινή μας συνεδρία έχουμε εδώ την Προεδρία της Μάλτας. Ε, εκπροσωπείται από τον ε, George Βέλα, που είναι ε, ο Υπουργός Εξωτερικών ε, της Μάλτας και είναι επίσης ε, ήταν και μέλος του κοινοβουλίου μας ε, κατά την προσκόρηση της Μάλτας και είχαμε συνεργαστεί και στην συμβατική συνέλευση για την Ευρώπη όταν συζητούσαμε για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ιστορικά πλέον γεγονότα. Χαιρόμαστε όλος ιδιαιτέρως ε, που είστε εδώ σήμερα. Ε, χαιρόμαστε πολύ που έχουμε εδώ μαζί μας την Μαλτέζικη Προεδρία. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε τα ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ξέρουμε, βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας ε, και βλέπουμε ε, κάθε φορά που εγώ είμαι εδώ στην Προεδρία της Συνεδρίασης μιλάμε για τις τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες που υπάρχουν και πόσο λίγοι είναι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχει ανθρωπιστική ανάγκη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, κρίση των προσφύγων ε, στην Ελλάδα, στις, ε, στην περιοχή των Βαλκανίων, έχουμε προβλήματα στο Νότιο Σουδάν, στη Συρία, στην Ιεμένη ε, και ανθρωπιστικές κρίσεις στην, ε, στις περιοχές αυτές. Είναι ένα θέμα λοιπόν που πιέζει την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως επίσης και ε, θέτει το πρόβλημα των πόρων που μπορούν να διατεθούν. Περιμένω λοιπόν εναγωνίω να ακούσω ποιε είναι οι δικέ σα προτεραιότητε και πώ θεωρείτε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι πολλαπλέ κρίσει και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ανακουφίσουμε τον ανθρώπινο πόνο και να ε, συνδέσουμε τον την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξική βοήθεια. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, μία ακόμη φορά να σας ε, ε, συγχαρώ επισήμως για την ε, εκλογή σας μία ακόμη φορά ως ε, Προέδρο αυτής της Επιτροπής αυτής. Πάρτε είναι πάρα πολύ σημαντικό που συζητούμε αυτή τη στιγμή που ε, πρέπει να συζητήσουμε ε, όλοι μαζί. Ε, κοντεύουμε στην 60η επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Μάλτα είναι το πιο μικρό μέλος, ένα μικρό νησί που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα όσα έχουν επιτευχθεί ε, σε αυτά τα τελευταία 60 χρόνια και να βεβαιωθούμε ότι θα βασιστούμε και θα δώσουμε, θα μεταλαμβαδεύσουμε στους πολίτες μας όλα τα θετικά αυτού του προγράμματος. Η Ευρώπη χρειάζεται μία νέα όθηση τώρα και οι πρόσφατες εξελίξεις ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δείξει την ανάγκη να έρθει πιο κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους πολίτες της και να ε, κοινωνήσει καλύτερα τα νέα μέτρα ε, να ώστε να έχουν οι πολίτες καλύτερες ευκαιρίες και να μπορούν οι πολίτες να επιτύχουν ε, όσο το δυνατόν περισσότερα σε σχέση με τις ανάγκες τους. Ε, τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν αφήσει σε όλους μας ε, σημάδια. Χρειάζεται ε, να αλλάξουμε πορεία, χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο κοντά στους πολίτες μας και έγιναν και γεγονότα, γεγονότα πέρσι που έχουν επηρεάσει την πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Μάλτα θέλει να συμμετέχει, να βάλει και εκείνη ε, το λιθαράκι της στην προσπάθεια αυτή. Ε, το Συμβούλιο σε συνεργασία με εσά θα είναι πραγματικά ε, καλύτερο. Θα καταφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ ε, πιο ισχυρή. Έξι μήνε είναι μικρό χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσουμε όμω να προχωρήσουμε με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Παράλληλα όμω είμαστε και ρεαλιστέ. Ξέρουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί μα, ξέρουμε ε, πού ε, βρίσκονται τα ισχυρά μα σημεία και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας ως ειλικρινείς συνομιλητές, χωρίς ε, μυστικά και θέλουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο σε ένα πνεύμα ειλικρίνειας ε, και με ανοιχτό πνεύμα. Ε, εμείς, ε, πολλά μέλη του Υπουργικού μας Συμβουλίου ήταν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο παρελθόν και ήταν και παρατηρητές πριν ε, η Μάλτα αποτελέσει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ε, το γεγονός ότι παραμείναμε στο Κοινοβούλιο μετά την προσχώρηση της Μάλτας μας βοήθησαν να καταλάβουμε τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπείται απευθείας τους Ευρωπαίους πολίτες. Είμαστε περήφανοι που παίρνουμε τα ενία της της ε, ε, Προεδρίας της ε, του Συμβουλίου σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα όθηση που θα σημαίνει ότι οι πολίτες θα προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον ως Ευρωπαίοι, ως καταναλωτές ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργάζονται μετανάστευση, ασφάλεια, ενιαία αγορά πολιτική γειτονίας, κοινωνική ένταξη και ε, θαλάσσια ε, θέματα. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ε, πολύ θεμητές ανησυχίες στον κόσμο που πρέπει να τις ακούσουμε. Δεν θα ήθελα να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες αυτές. Ε, θα αναφερθώ μόνο ε, στο πρόγραμμά μας όσον αφορά το θέμα με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή σας και ε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας ε, για να συζητήσω το θέμα αυτό ε, η Προεδρία της ε, Μάλτας, ε, οι προτεραιότητες της Προεδρίας μας για τον ανθρωπιστικό τομέα, δεδομένων των εργασιών που έχουν ήδη έχουν δρομολογηθεί και στο Κοινοβούλιο και στη δική σας Επιτροπή, έχουν αυτήν την κοινή ανησυχία που είναι η ανθρωπιστική, τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Συνεργαζόμαστε με τους Ολλανδούς και Σλοβάκους εταίρους μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ε, συμπεφωνημένους στόχους του ε, προγράμματος ε, του του, του, του προγράμματος του τρίο και θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί εξασφαλίσατε μια πολύ ομαλή μετάβαση στη δική μας Προεδρία και κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρία μας θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την πρόοδο ε, των, ε, που έχουν σημειώσει προηγούμενες Προεδρίες όσο καλύτερα μπορούμε ε, η παγκόσμια ανθρωπιστική κατάσταση βέβαια και είμαι επίοικης όταν το λέω αυτό, όχι σε πολύ καλή κατάσταση. Η τελευταία παγκόσμια ανθρωπιστική επισκόπηση για το 2015, ε, ο, ο συντονιστής για τα θέματα αυτό, Στίβεν Ομπράιαν, είπε ότι η εμβέλεια της ανθρωπιστικής κρίσης είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τότε που ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν ε, υπάρχει ε, στη μνήμη μας, ε, δεν έχει ξαναυπάρξει μια κατάσταση κατά την οποία να χρειάζεται τόσο πολύ αλληλεγγύη για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει στην αξιοπρέπεια. Σε 93, εκατομμύρια είναι τα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη, πάνω από 128 εκατομμύρια άτομα ε, πλήττονται από ε, ε, εκτοπισμό, είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα φτώχειας. Είναι λοιπόν μια τεράστια ανθρωπιστική ε, κρίση που θα απαιτήσει 22,5 δισεκατομμύρια ε, για να ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα 193 άτομα, εκατομμύρια άτομα που χρειάζονται τόσο πολύ την βοήθειά μας. Υπάρχει εκτοπισμός εντός των χωρών αλλά και διασυνοριακά. Υπάρχουν προβλήματα, φαινόμενα όπως το Ελνίνιο, πλημμύρες, θεομηνίες που που ε, απειλούν την επιβίωση κάποιων ευάλωτων ομάδων. Επομένως, η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανάπτυξη νέων ανθρωπιστικών ε, εργαλείων είναι πιο απαραίτητα από ποτέ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνεισφορά, είναι αδύνατον να ακολουθήσει κανείς το ρυθμό της αύξησης των ανθρωπιστικών αναγκών. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα ε, που καταγράφηκε στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο πέρσι Προσπαθούμε να έχουμε ένα σύστημα πιο αποδοτικό, πιο προβλέψιμο και πιο ευέλικτο. Δεν είναι δυνατόν η ανθρωπιστική βοήθεια μόνη της να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ε, τα περισσότερα προβλήματα που είναι πιο ευάλωτοι. Και αυτό ε, αποκρισταλώθηκε σε τρεις προτεραιότητες. Οι βασικές αιτίες που οδηγούν σε τεράστιες ροές προσφύγων και εκτοπισμένων, ε, πρόληψη και ε, ε, πρόληψη των ε, συγκρούσεων και όπως επίσης, όπως επίσης και ανάπτυξη ανθρωπιστικών, ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, εμείς έχουμε σκοπό να συνεισφέρουμε σε μια βελτιωμένη και πιο συντονισμένη ανθρωπιστική βοήθεια, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συγκρούσεις που συντελούνται εδώ και μεγάλο, που μένονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί ε, και η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Ε, θέλουμε να είμαστε υπέρμαχοι ε, των ανθρωπιστικών της ανθρωπιστικής προσέγγισης ε, στις χώρες όπου δεν είναι επαρκής αυτή ε, και ειδικότερα θέλουμε να προστατεύσουμε τις πιο, τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Θέλουμε λοιπόν να εντοπίσουμε τρόπους να βελτιώσουμε το ευρύτερο ανθρωπιστικό σύστημα και να προωθήσουμε μια συνεπή συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών μετά από τις καταστροφές. Ε, στο πλαίσιο ε, αυτού του ευρύτερου στόχου έχουμε το ανθρωπιστικό μας θεματολόγιο μετά από την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο. Ε, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες αλλά και συλλογικές προτεραιότητες για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ανθρώπινο πόνο παντού σε όλο τον κόσμο. Ε, αυτό θα το κάνουμε βέβαια με τους ε, εταίρους μας και μίας ε, πλατφόρμας την οποία έχει δημιουργήσει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων. Προσπαθούν λοιπόν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου για να εξασφαλίσουμε ότι σε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει κατάλληλη παρακολούθηση και ένας μηχανισμός υποβολής εκθέσεων ως προς τις δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, το Μάιο για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο. Ε, θέλουμε λοιπόν να υπάρξει σε παγκόσμιο επίπεδο συμπληρωματικότητα και συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και σε σχέση με την πολιτική που αποφασίστηκε στη Σύνοδο. Ε, οι δεσμεύσει των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο και οι τρεις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Συνένεση στην Ανθρωπιστική ε, βοήθεια ε, θα αποτελέσουν τμήμα της δεύτερης βασικής μας προτεραιότητας που είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την ανθρωπιστική αρρωγή. Πράγματι, η συνένεση αυτή επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες για να ε, ενισχύσει τις ανθρωπιστικές δράσεις και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, την τήρηση ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μια προσέγγιση βάση στοιχείων και ενισχυμένο συντονισμό. Η Προεδρία θα εξασφαλίσει ότι οι τρεις αυτές προτεραιότητες βάσει του σχεδίου δράσης που, έχει αποφασιστεί σε, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα. Ιδίως ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί στην συνδιάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά την, ε, ε, εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει εκπονηθεί θα προσπαθήσουμε να διαδραματίσουμε έναν ενεργό ρόλο προκειμένου να ευξήσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας υποστηρίζοντας την εκπλήρωση ε, του δεύτερου σχεδίου υλοποίησης. Η ο δεύτερος στόχος της Μαλτέζικης Προεδρίας θα είναι η προσπάθεια ανάπτυξης του ε, κόμβου ανθρωπιστικής βοήθειας. Πολλές φορές η, ε, τα όρια μεταξύ ε, αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας είναι θολά. Ακριβώς λόγω της περιπλοκότητας των καταστάσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας, βραχυχρόνιας άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας. Στόχος μας είναι να γεβηρωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Ιδιαίτερη προσοχή θέλουμε να δώσουμε και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας ε, ε, και της αντοχής των εκτοπισμένων ε, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω. Όσον αφορά τους αναγκαστικά εκτοπισμένους η Προεδρία ε, θα προσπαθήσει να αναπτύξει, να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα με θεματικά και γεωγραφικά παραδείγματα ε, αντιμετώπισης του προβλήματος αυτούς και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 65 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν πλέον εκτοπισμένοι, κάτι που ε, ε, που προκαλεί ε, ένα μακροχρόνιο πρόβλημα θα προσπαθήσουμε να βρούμε βιώσιμες λύσεις για τους ε, πληγέντες πληθυσμούς συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων και εκείνων που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Η Προεδρία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανθρωπιστικές προκλήσεις ε, τονίζοντας τα τροτά σημεία και τις ανάγκες τόσο των μεταναστών όσο και των κοινοτήτων και των χωρών που τις υποδέχονται. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η προστασία ε, των ε, πληθυσμών. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πολλές φορές παραγνωρίζεται στις ε, ένοπλες συγκρούσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. Υπάρχουν στοχευμένες επιθέσεις σε αμάχους, υπάρχει καταστροφή ανθρωπιστικών και ιατρικών εγκαταστάσεων, ε, ε, υποδομών κοινής ωφέλειας η Προεδρία μας λοιπόν θα προσπαθήσει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανθρωπιστική προστασία τόσο εντός όσο και πέραν του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Άλλες προτεραιότητες. Διατροφή και επιστημιστική ασφάλεια. Θα εξασφαλίσουμε να παραμείνει αυτό ο τομέας ένα σημαντικό θέμα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Συνεργασία μεταξύ ε, αρχών ε, πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ των ε, διαφόρων φορέων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η Προεδρία της Μάλτας είναι στοχοπροσιλωμένη, γνωρίζει και έχει επίγνωση τις ευθύνες της σχετικά με την, με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς εκείνους που το χρειάζονται. Προσβλέπουμε λοιπόν με ε, μεγάλη χαρά προκειμένου να καταστήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια πιο αποτελεσματική και πιο ολοκληρωμένη. Στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας μας προσβλέπουμε στη συνεργασία με εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσίαση αυτή. Φαίνεται ότι έχετε φορτωμένο πρόγραμμα ε, τα, τους επόμενους έξι μήνες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τρεις ομιλητές έχουμε αυτή τη στιγμή στον κατάλογο. Ε, αν θέλετε και εσείς το λόγο, παρακαλώ, ε, κάντε μας ένα νόημα για να σας καταγράψουμε. Ξεκινούμε. Με τον Ερήγη Σαλόμ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τη Λίντα και τα άλλα μέλη της Προεδρίας, ε, να τους συγχαρώ για την εκλογή τους σήμερα το πρωί και ε, ευελπιστώ βεβαίως ότι θα συνεχίσουμε τα επόμενα δυόμιση χρόνια να συνεργαζόμαστε αρμονικά. Δεύτερον και σημαντικό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό και κυρίως τη Μάλτα για τον ρόλο τον οποίο έχει παίξει όσον αφορά θέματα τα οποία σχετίζονται με την μετανάστευση, με την ανθρωπιστική κρίση, με τους ε, ε, πρόσφυγες ε, διότι για τα θέματα αυτά ε, πραγματικά η Βαλέτα αποτελεί παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων και βεβαίως αποτελεί και σημείο αναφοράς όσον αφορά τις οικονομικές συμφωνίες και την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αυτό. Ο Υπουργός ξεκίνησε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρείται και θεωρείται ακόμα ως πρότυπο. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι όχι μονάχα θεωρείται σαν ένα συνολικό ε, σχέδιο ή πρόγραμμα, αλλά και ειδικά σε θέματα ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως πρέπει να πούμε ότι ένα από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι είναι απομακρυσμένοι από, τις, από τους πολίτες και πρέπει να τους πλησιάζει περισσότερο ε, και νομίζω ότι μέσω της ε, ανθρωπιστικής δράσης υπάρχουν πολίτες που βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια, πολύ πιο κοντά λέω από ότι οι κυβερνήσεις των κρατών η κοινωνία, οι μικρές κοινότητες ε, προχωράνε περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη ε, συνειδητοποίηση της ε, κατάστασης και των προβλημάτων ή πολύ περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, συνειδητοποιούν τα προβλήματα από ότι η πλειοψηφία, ας πούμε, των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το να είναι κανείς κοντά στους ε, πολίτες ε, σημαίνει να είναι και ευαίσθητος σε αυτήν την θέση της, των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που που αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα το ότι έχει εκλεγεί πρόεδρος ας πούμε μίας ε, χώρας ένας άνθρωπος ο οποίος ε, θα την μετατρέψει σε δεύτερη ε, δύναμη στον κόσμο μέσα από πολιτικές, εμπορικές κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά την ανάπτυξη και την και την ανθρωπιστική βοήθεια θα δώσει σε αυτά λιγότερη σημασία. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσουμε από κοντά ε, την ε, ε, ε, παγκόσμια διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει οπωσδήποτε όσο γίνεται πιο γρήγορα να εγκαθιδρύσουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και κατά πόσο να αντιμετωπίζουμε τις υποχρεώσεις μας και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως μεμονωμένα με μονομένα ε, κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να γίνει στην ε, διάσκεψη της ε, Κωνσταντίνου Πόλεως. Ανάπτυξη λοιπόν του σχεδίου δράσεως ε, και όσον αφορά την ε, διασύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ανθρωπιστική ε, δράση. Το έχουμε πει πολλές φορές και το υπογραμμίζω γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Υπουργό. Είναι απαραίτητο μεταξύ των μελών της Επιτροπής, βεβαίως τα γνωρίζουμε, αλλά είναι σημαντικό να τα ξαναπούμε, ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις έχουν πλέον μεγαλύτερη διάρκεια. Δυστυχώς εγκαθίστανται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αρκεί η άμεση βοήθεια, δεν αρκεί η βράχη πρόθεσμη βοήθεια είναι απαραίτητες και άλλες δράσεις. Η εκπαίδευση, όπως είπατε, η ιατρική ε, αρρωγή, έτσι ώστε μετά από την πρώτη ανταπόκριση σε μια ανθρωπιστική κρίση να εγκατασταθεί και αυτή η διαρκής και ανθεκτική βοήθεια. Όσον αφορά την προστασία των πληθυσμών, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο βεβαίως που είναι πολύ σημαντικό είναι να προστατευθεί ε, η κοινότητα, ο πληθυσμός ο οποίος ε, διανύει ανθρωπιστική κρίση. Ωστόσο θα πρέπει να ε, προστατεύουμε και τους, ε, σε όσους συμμετέχουν, σε αυτούς που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίοι σφαγιάζονται, οι οποίοι δολοφονούνται, χάνουν τη ζωή τους μέσα σε σκηνές, μέσα σε νοσοκομεία, ε, μέσα σε κέντρα βοήθειας. Το έχουμε πει, το έχουμε πει αυτό. Ε, και βέβαια όλα αυτά που αναφέρονται στις συνήθεις εκθέσεις και της Κομισιόν και της δικές μας σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης κλπ. Αυτά είναι σταθερά. Ε, δεν θα πω πολλά πράγματα ακόμα, αλλά πρέπει να πω ότι φυσικά θα πρέπει να δούμε και την ανθρωπιστική ανάγκη που βρίσκεται εκτός των συνόρων μας στα σύνορά μας έχουμε ένα εκατομμύριο, ενάμιση εκατομμύριο ανθρώπους, τους οποίους βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε, να προστατέψουμε, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο έχουμε 60-70 εκατομμύρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Να μην λησμονούμε την σχετικότητα, το, το σχετικό μέγεθος των προβλημάτων. Πάντως, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες ε, ε, είδαμε, διανύσαμε, ζήσαμε πραγματικές ε, ε, πραγματικές καταστάσεις επίγουσες στη Σερβία, στην Ελλάδα, ε, στη Τσεχική Δημοκρατία και σε άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του ψύχους ιδιαίτερος. Επομένως η Μαλτέζικη Προεδρία περιμένουμε να πιέσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να έχουν ένα μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα αντιμετώπισης του χειμώνα. Γιατί είδαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο καιρό. Πέρα σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αναφέρει η Προεδρία, εγώ θα ζητούσα σε ορισμένα σημεία να συμπεριλάβει περισσότερο και τη διάσταση του φύλου και της ηλικίας. Ε, γιατί ξέρουμε ότι και οι ηλικιωμένοι και τα νέα παιδιά, σε, τα μικρά παιδιά ε, σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης ε, αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και το φύλλο επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά τώρα την καταπολέμηση των υποχρεωτικών εκτοπισμών, υπάρχει ανακοίνωση της Κομισιόν ε, τον Απρίλιο, του Απριλίου μάλλον του 2016, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή. Σε αυτήν την ε, ανακοίνωση λοιπόν υπήρχαν διάφορα θετικά στοιχεία, όμως ούτε εγώ ο ίδιος ούτε και η ομάδα μου βλέπω διασύνδεση μεταξύ του περιεχομένου της ανακοίνωσης και των προτεραιοτήτων της Προεδρίας. Ε, θα ήθελα πάντως να συγχαρώ την Μάλτα επί τη αναλήψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευελπιστώ ότι θα μεταλαμπαδεύσει και σε όλους μας αυτήν την υπερηφάνεια ε, και το στένος αυτής της μικρής ε, χώρας. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Στρασβούργου ο, κύριος ο πρόεδρος είπε ότι Χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκε η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γιατί πλέον ε, το Λουξεμβούργο ε, μπορεί να μην γινόταν πλέον να έχανε τη θέση ως η μικρότερη χώρα τουλάχιστον δεν ήταν η μόνη πολύ μικρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω ε, έχοντας ε, συνεργαστεί και με, την, ε, και με εσάς και με τη Μαλτέζικη Προεδρία και στη μεσάς διάσκεψη των Προέδρων γνωρίζω πάρα πολύ καλά την δυνατότητα καλής λειτουργίας της Μάλτας και στα πλαίσια της Προεδρίας. Σας συγχαίρω λοιπόν επί την αλήψη σας καθηκόντων. Θα είμαστε πάντα κοντά σας και θα σας υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Ενρίκε, Μπόγκταν και με τον Νόρμπερτ Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστούμε πολύ για την λεπτομερή ε, παρουσίαση των στόχων της Προεδρίας και όχι μονάχα σχετικά και αποκλειστικά με την ανθρωπιστική κρίση γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να ιδωθεί και από μια ευρύτερη ε, σκοπιά. Θα συμφωνήσω με όλα ε, όσα είπε ο προλαλής σας ε, συνάδελφος και να πω ότι βλέποντας, βλέποντας το χάρτη του κόσμου ε, υπάρχει μια, ένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται τεχνικό. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με την ισπανική διαρμηνία. Ε, εγώ ακούω, λέει η συνάδελφος Ισπανικά, μάλλον δεν έχεις βάλει τα σωστά ακουστικά, Ενρίκε. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε λίγο τον χάρτη του κόσμου και ε, να δούμε λίγο τα κέντρα της ανθρωπιστικής κρίσης σε αυτόν τον κόσμο. 90% ε, αυτών των καταστάσεων κρίσης ε, βρίσκεται στην Αφρική και τα, σε μεγάλο ποσοστό αφορά γυναίκες και παιδιά. Ε, και ε, συνήθως όταν μιλάμε για νέους αναφερόμαστε σε ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Προκύπτει λοιπόν η ερώτηση. Η Προεδρία πιστεύει ότι είναι δυνατόν να ε, ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους που είναι ιδιαίτερος ευαίσθητοι. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νόιζα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και σας ευχαριστώ και για το γεγονός ότι και στο προηγούμενο εξάμεινο κατά τη φάση της ε, προετοιμασίας της Προεδρίας σας εργαστήκατε σκληρά. Ε, έχετε αναλάβει ένα τιτάνιο έργο παρά, το μικρό μέγεθος της χώρας σας αλλά από την εμπειρία μου με τους συναδέλφους σας και τους συνεργάτες σας μπορώ να σας πω και εγώ ότι είστε άριστα προετοιμασμένοι για την Προεδρία. Γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι θα επιτύχετε και αυτούς τους υψηλούς στόχους που έχετε θέσει. Είπατε ότι, ε, έχετε, ότι είστε μια φιλοευρωπαϊκή ε, κυβέρνηση με πολλά μέλη της να έχουν ε, θητεύσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό ε, αν συνέβαινε και σε άλλες χώρες ενδεχομένως ε, θα είχαμε αποφύγει διάφορα προβλήματα. Ως ε, μικρή νησιωτική χώρα έχετε βιώσει με ιδιαίτερη ένταση τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε και αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμη αρρωγή, αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των ανθρώπων. Δεν ε, έχετε δίκιο, δεν πρέπει να συγχέονται οι δύο αυτές ε, μορφές της βοήθειας, της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής αλλά θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο εντός της οποίας θα παρέχεται η κάθε μία. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει με επιτακτικότητα να αντιμετωπίσετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα Βαλκάνια. Την, ε, στην τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο συζητήσαμε το θέμα αυτό και καταλήξαμε ε, ε, στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση είναι πλέον απάνθρωπη εκεί. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να αναλυφθεί η δράση σε συνεργασία και με τις χώρες των Βαλκανίων ε, και σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των προσφύγων εκεί. Ε, ένα ακόμη θέμα ε, θα ήθελα να αναφέρω. Συνένεση όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Στον τομέα αυτό η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Αν έχουμε αυτό στο επίκεντρο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε γρήγορα να καταλήξουμε σε συμφωνία στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου προκειμένου στη ε, συνέχεια ε, να καταλήξουμε σε ένα καλό ε, αποτέλεσμα τον Ιούνιο στην Μάλτα, στην διάσκεψη που οργανώνεται. Τέλος, χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι λάβατε υπόψη σας τις, να ε, ε, διοργανωθεί η διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ACP στην Μάλτα ακριβώς γιατί είναι σημαντικό εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλουμε θετικά μηνύματα προς τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ ο Σαλ Γκόρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ τη μόνη ε, χώρα που ε, ευνοήθηκε από την, ε, προ... από την προσχώρηση της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εγώ πραγματικά δεν έχω καμία αμφιβολία για την πρόθεσή σας να σημειωθεί πρόοδος το... Υπάρχουν κάποιες, υπάρχει χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική κρίση, υπάρχουν κάποια προβλήματα που τα γνωρίζουμε ήδη και υπάρχουν και τα ε, προβλήματα με τους πρόσφυγες. Και αυτό που είναι έτσι μια, κό, μια ε, κόκκινη γραμμή που φαίνεται ε, είναι πραγματικά η ανεπάρκεια των πόρων. Οι λόγοι της ανεπάρκειας αυτής έχει να κάνει με την άρνηση ορισμένων ορισμένων χωρών να αντεπεξέλθουν σε κάποιους στόχους οποίους είχαν προσυπογράψει. Κάτι ακόμη θα ήθελα να παρατηρήσω, η ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας. Τι το ιδιαίτερο έχει, είναι η ουδετερότητά της και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε ε, με νύχια και με δόντια, δεν πρέπει να αφήσουμε να πλανάται η παραμικρή αμφιβολία σε σχέση με την ιδιαιτερότητα αυτή, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα, χωρίς καμία απολύτως ε, δυσκολία, ε, μαζί με άλλους ε, εταίρους που βοηθούν ε, στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, μπορούμε να βγούμε από τις επιταγές της Realpolitik. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι την ουδετερότητα. Και αυτή η ουδετερότητα με οδηγεί στην τρίτη μου παρατήρηση. Και η τρίτη μου παρατήρηση αφορά ένα θεσμικό ζήτημα. Βρίσκω αρκετά περίεργο το ότι η Προεδρία ε, του ε, Συμβουλίου, μας, βλέπει, μας συναντά ανεπίσημα για να μιλήσουμε για την ανάπτυξη, αλλά ε, στην ολομέλεια της ε, Επιτροπής μας δεν μπορούμε να συζητήσουμε μόνο με ανθρωπιστικά ζητήματα, που δεν λέω ότι είναι απλό ζήτημα, αλλά πάση περιπτώσει μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. όσον αφορά λοιπόν την σε προεδρία, ο βασικός στόχος της είναι να συντονίζει ε, τον νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, από απόψεως ε, νομοθετικής έχουμε πολλά να κάνουμε, ε, αλλά ε, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτε άλλο εκτός από την Ευρωπαϊκή Συνένεση για τα ανθρωπιστικά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, δεν, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Υπουργοί Εξωτερικών μπορούν να έρθουν και να μιλήσουν στην Επιτροπή Ανάπτυξης ή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά μπορούμε για τα θέματα της ανάπτυξης να μιλούμε μόνο επισήμω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω από, ε, καθόλου. Ε, εγώ ε, δεν λέω ότι Πιστεύω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε με την ε, κυρία ε, ε, Μογκερίνη. Δεν λέω βέβαια ότι δεν έχει έρθει πολλέ φορέ, ούτε έχω καμία αμφιβολία για την διαθεσιμότητά τη και τι καλέ τη προθέσει. Όμω νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θέσουμε. Το θέμα αυτή τη νομοθετική πρόοδου, του συντονισμού που πρέπει να γίνει μεταξύ των 28, ε, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συστηματική προσέγγιση και αναφέρομαι στην χρηματοδότηση. Ε, το πρόβλημα της χρηματοδότησης πρέπει να το συζητήσουμε. Ε, ποιος ζητάει το λόγο από τα κράτη-μέλη που αρνήθηκαν να, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Κανένας. Κανένας δεν του ζήτησε το λόγο. Κάθε φορά το λέω, κανένα δεν μου απαντάει. Εφτά χρόνια ε, το θέτουμε αυτό το θέμα και δεν υπάρχει καμία συνέχεια. Και δεν το λέω σε σας προσωπικά, αλλά σας κάνω εσάς προσωπικά μία έκκληση για να μπορέσετε να το μεταφέρετε αυτό στα θεσμικά ε, βήματα στα οποία έχετε πρόσβαση, ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτόν τον παραλογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Χάιντι Χάουταλα. Για τώρα και συνέχεια θα κάνουμε έναν ακόμη γύρο ερωτήσεων. Ε, μιλάμε για μια ανθρωπιστική ε, κρίση, για μια ε, κατάσταση η οποία είναι πολύ σοβαρή και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν πρόκειται να λήξει γρήγορα. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι χθες στο Ελσίνκι ολοκληρώθηκε μία μεγάλη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών ε, που ασχολήθηκε με την ανθρωπιστική κρίση στην Συρία καθώς επίσης ε, και την βοήθεια που χρειάζεται η Συρία. Ο Φίλιππο Γκράντι από πλευράς ε, υπεύθυνος για τους για τους πρόσφυγες ε, ε, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι χρειάζονται τέσσερα δις ε, για να βοηθηθούν αποτελεσματικά γιατί θα υπάρξουν περίπου 4,5 ακόμα εκατομμύρια Σύριοι οι οποίοι θα φύγουν από την χώρα τους. Αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Επίσης ακούσαμε πολλά ε, και για την Συρία όπου λείπουν, ε, έχουν ανάγκη από γιατρούς, ε, από φαρμακευτικό υλικό. Ξέρετε ότι ε, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο, από άλλες ε, ασθένειες, διότι δεν έχουν πρόσβαση στην ε, ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Σε μερικές περιπτώσεις ένας γιατρός είναι υπεύθυνος για 4 και 5.000 ανθρώπους. Ε, τι θα κάνετε λοιπόν για να βοηθήσετε επιτόπου στη Συρία, ε, ε, τι θα κάνετε για να βοηθήσετε και τις πιο ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, κυρίως γυναίκες και νεαρές κοπέλες. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Λίτς και Έλλης Σνάιτ στον επόμενο γύρο. Τελειώσαμε προς το παρόν με τον πρώτο γύρο. Τερέσα, ποιος άλλος θέλει το λόγο. Απλά τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ξεκινώντας με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Ε, συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν και ε, με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε τα ζητήματα των συναισθηματικά φορτισμένο. Και εμείς φυσικά έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Είπατε ε, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επανέλθει κοντά στους πολίτες της. Πράγματι, έχουν υπάρξει διάφορες ε, εξελίξεις, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια ε, και είναι δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και αυτό ε, ε, αντικατοπτρίζεται και στην άνοδο διαφόρων πολιτικών ρευμάτων που ε, έχει πάρει στα τελευταία χρόνια. Ε, εμείς με ειλικρίνεια πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την παρέμβασή της σε όλους τους τομείς. Είπατε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Εκτός από το γεγονός ότι στην σχετική συνδιάσκεψη υπήρχε συμμετοχή υψηλού επίπεδου, ε, υπήρξαν ε, ε, πάνω από 3.000 δεσμεύσεις έκτοτε και από την Κωνσταντινούπολη και έπειτα. Εμείς λοιπόν είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων και ότι δεν θα υπάρξει επαναχώρηση από τις χώρες που έχουν αναλάβει τις δεσμεύσεις αυτές. Γι' αυτό και ε, έχουμε δημιουργήσει την διαδικτυακή πλατφόρμα προκειμένου να παρακολουθείτε η πρόοδος. Όσον αφορά την ε, ανθρωπιστική ε, κρίση, την προσφυγική κρίση, θεωρώ δεδομένο ότι δεν διαφωνούμε επί της ουσίας σε κάτι. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται 22 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τους εκατομμύρια εκτοπισμένους που υπάρχουν φέτος. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι ε, πρέπει να ε, μην χάνουμε από τον ε, προσανατολισμό στο γεγονός ότι υπάρχουν και ε, ε, κρίσεις οι οποίες ε, έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια και δεν είναι απλά βραχυχρόνιες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επίγνωση ότι οτιδήποτε ε, χορηγούμε, οτιδήποτε ε, δαπανούμε ως ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να έχει και τα ε, επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητάτε και εσείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή πολύ συχνά. Και δεν υπάρχει μόνο η αλτρουιστική διάσταση αυτού του θέματος, ε, το δικαίωμα δηλαδή των ε, ανθρώπων ένα, ε, σε μια αξιοπρεπή εκπαίδευση είναι και ζήτημα ζωής και θανάτου πολλές φορές, καθώς ε, η εκπαίδευση μπορεί να γλιτώσει παιδιά από την παιδική πορνεία, από την αναγκαστική ε, εργασία, από το ε, οργανωμένο έγκλημα. Επομένως, είναι και ένα μέσο για την πρόληψη και την αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον. Είναι θετικό λοιπόν το γεγονός ότι ε, η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών που πλήττονται από κρίσεις ε, στον ένα ή στον άλλο βαθμό ε, έχει πρόσβαση σε ορισμένες δομές εκπαίδευσης. Αυτό είναι και ο σημαντικότερος στόχος. Είναι πρόκληση γιατί δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι εκείνοι που θέλουν να παρέχουν εκπαίδευση μπορούν και να έχουν πρόσβαση στα παιδιά. Είδαμε ότι ακόμη και η ιατρική βοήθεια πολλές φορές στη Συρία δεν μπορούσε να φτάσει στο στόχο της. Αναφέρατε επίσης ε, αναφερθήκατε επίσης ε, στην ε, ε, ε, στην έντονη ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες ε, στον, στα, Βαλ, στα Βαλκάνια. Αναφερθήκατε στην ανάγκη παρακολούθησης των ανθρώπων αυτών Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, ε, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι αποτελεί μία από τις προτεραιότητες μας και πρέπει να σας πω ότι στη Μάλτα έχουμε από τις πλέον προηγμένες νομοθεσίες όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Ε, τα τελευταία τρία χρόνια κάναμε πολύ ε, γρήγορη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανθρωπιστικής διάσκεψης. Ταυτόχρονα, στη διάρκεια της Προεδρίας θα διοργανώσουμε στη Μάλτα δύο εκδηλώσεις. Μία κατά της βία ε, κατά των γυναικών και υψηλού επίπεδου ε, η, υπουργική διάσκεψη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι μα απασχολούν αυτά τα ζητήματα και ε, εγώ εδώ ε, ήρθα βεβαίως απλώς για να σας ε, παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ζητήματα τρίτης ηλικίας. Μετανάστες και πρόσφυγες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στο πρόγραμμα της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας έχουν ληφθεί υπόψη όλα αυτά Για τα μέτρα για το χειμώνα. Προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να ε, επιτύχουμε μια μορφή αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης. Δεν θέλω να μπω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες γιατί ανοίγονται πολλά θέματα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και που επιδιώκουμε να καταφέρουμε είναι με κάποιον τρόπο να αμβλύνουμε τις, τις ε, τεράστιες διαφορές ε, απόψεων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών ε, να αμβλύνουμε λέω, δεν λέω ότι θα γεφυρώσουμε το χάσμα πλήρως Έχουμε σε κάθε περίπτωση εξετάσει τις απόψεις και τις γνώμες που έχουν εκφράσει επικεφαλής κυβερνήσεων ε, και επιδιώκουμε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμβιβάσουμε προς όφελος όλων όσο γίνεται τις διαφορετικές απόψεις είπατε επίσης για τους ε, αναγκαστικά εκτοπισμένους ε, και δεν υπάρχει βεβαίως αμφιβολία ότι είναι και αυτό ένα πολύ σοβαρό ζήτημα καθώς ε, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έχουν επιτακτική ανάγκη να λάβουν βοήθεια. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην Κοχάφα και εγώ γνωρίζω ε, ότι ε, λόγω της, κατα... της θέσης, της γεωγραφικής θέσης της ε, χώρας μου είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και τις δύο οπτικές και την οπτική της Ευρώπης και την οπτική των Αφρικανικών κρατών. Έχουμε εμπειρία από τις εμπειρίες, έχουμε εμπειρίες από τις σχέσεις μας με Αφρικανικές χώρες και μπορώ να σας πω ότι είμαστε αρκετά προσεκτικοί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλούμε για την Αφρική λες και είναι μια, λες και είναι μια χώρα. Πρόκειται μια τεράστια Ήπειρο και ε, Ήπειρος της οποίας ο πληθυσμός στο άμεσο μέλλον θα αυξηθεί ε, εκθετικά ε, και βεβαίως η δημογραφική αυτή έκρηξη ε, μπορεί να δημιουργήσει και μελλοντικά διάφορα προβλήματα. Επίσης γυναίκες και παιδιά στη θεματολογία αυτή, ιδίω γυναίκες παιδιά ως πρόσφυγες, οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια, πιστεύω ότι οι αρχές ε, που χρησιμοποιούμε, που εφαρμόζουμε ε, ε, συστηματικά, ε, όσον αφορά τη, την, τις γυναίκες και τα παιδιά ισχύουν ακόμη περισσότερο της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης, της ε, ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ε, φυσικά ισχύει και για τους άνδρες, ισχύουν αυτές οι αρχές και για τους άνδρες, αλλά ιδίω για τα παιδιά και τις γυναίκες, τις εγγύους πολλές φορές ε, ή τις μητέρες μικρών παιδιών, οι αρχές αυτές έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ακριβώς γιατί ακόμη και από τα στοιχεία μας προκύπτει ότι ο αριθμός και το ποσοστό των ε, παιδιών που καταφτάνουν στην Ευρώπη ως μετανάστες δεν αντιστοιχεί ε, πάντοτε με τον συνολικό αριθμό ε, των προσφύγων που καταφτάνουν στην Ευρώπη. Αν δείτε ε, δηλαδή τους αριθμούς των μεταναστών και προσφύγων που καταφθάνουν στην Ιταλία από τη Σενεγάλη, από άλλες αφρικανικές χώρες, ε, έρχονται από συγκεκριμένα ε, ομάδα χωρών, Ερυθρέα και Τα παιδιά όμως, τα παιδιά μετανάστες πολλές φορές έρχονται, προέρχονται από άλλες χώρες. Αυτό είναι μια πηγή ανησυχία πολύ μεγάλη για εμά, ακριβώ γιατί καταδεικνύει ότι ενδεχομένω τα παιδιά αυτά είναι ε, αντικείμενα ε, εμπορία, ελαφρέα εμπορία ανθρώπων. Ε, άλλωστε γνωρίζουμε όλοι ότι χιλιάδες παιδιά έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεχομένως να είναι λοιπόν θύματα ε, διακίνησης ανθρώπων, ε, παιδικής ε, πορνείας, καταναγκαστικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα παρέχουμε στους, στα παιδιά αυτά δυνατότητες και ευκαιρίες μιας καλύτερης ζωής και γνωρίζω ότι ετοιμάζεται στην Επιτροπή σας και ένα σχετικό ψήφισμα ε, για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αναφέρομαι ε, κυρίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται από τη Μέση Ανατολή είναι πράγματι πρόσφυγες που, που συνδέεται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται πράγματι με την εμπόλεμη κατάσταση της Συρίας και οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως ε, πιέζουν σημαντικά τον Λίβανο, την Ιορδανία και μέχρι και την ε, συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και την χώρα αυτή και από εκεί βεβαίως και τις ε, χώρες κεντρικής Ευρώπης. Κύριε Νόισερ, κάνετε μια πολύ σημαντική παρατήρηση ότι ε, χρειάζονται και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά χρειάζονται και μακροπρόθεσμα σχέδια. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που είπατε, ακριβώς γιατί αυτές αυτή η κρίση ε, ενδεχομένως να τραβήξει σε πολύ μεγάλο μάκρος χρονικό και αυτό αφορά την Ευρώπη ολόκληρο, γιατί, ε, ολόκληρη, γιατί ελπίζουμε κάποια στιγμή η κατάσταση στη Συρία να διευθετηθεί. Πολλοί εκτοπισμένοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Το πρόβλημα της Αφρικής όμως δεν πρόκειται να λυθεί τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Πρόκειται για μετανάστες και όχι για πρόσφυγες. Ε, επομένως πρέπει εκ των προτέρων να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τα επόμενα 20-25 χρόνια ε, οπότε και αναμένεται αυτή η δημογραφική έκρηξη στην Αφρική. Αναφερθήκατε επίσης και στα μέτρα για το χειμώνα, ε, για τους πρόσφυγες ε, στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο της συνέννησης για την ανάπτυξη, ε, έχουμε μιλήσει και στο γεύμα για αυτό το θέμα, υπάρχει σε κάθε περίπτωση Επιδίωξε από την πλευρά μας ως Προεδρίας να καταλήξουμε με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατό σε ένα κείμενο ε, ώστε μέχρι το τέλος του εξαμήνου να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας. Αν δεν τα καταφέρουμε βεβαίως θα δώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου. Ε, επίσης ε, ε ε, ξανατονίζω ότι η συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ θα γίνει στην ε, ε, Μάλτα τον Ιούνιο έπειτα από δικές σας παρενέσεις και παροτρύνσεις. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η συνδιάσκεψη αυτή θα στεφθεί με επιτυχία. Τα οργανωτικά στοιχεία έχουν ήδη οριστικοποιηθεί ε, ελπίζω λοιπόν να στεφτεί με επιτυχία. Κύριε Γκιόρενς, μιλήσατε για τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται φυσικά για την ε, πρόκληση που αντιμετωπίζουν ε, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι λίγες ευρωπαϊκές χώρες που επομίζονται αυτή την ευθύνη την ευθύνη δηλαδή πως πολιτισμένες και δημοκρατικές χώρες αντιμετωπίζουμε. Δεν θα σας δώσω στοιχεία γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ε, πολλές δεσμεύσεις ε, αναλαμβάνονται. Παρ' όλα αυτά... Σε κάθε περίπτωση αυτό που ε, πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ε, η συμβολή όλων των κρατών μελών δεν θα είναι ε, για μία και μόνο φορά. Χρειάζεται μία σε βάθος χρόνου διαχείριση της κατάστασης και βεβαίως αποτελεί στόχο μας να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια κάποια ευελιξία όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των ε, κονδυλίων ε, και την ε, άρση ενδεχομένως ορισμένων πολύ αυστηρών κανόνων που σχετίζονται με αυτήν, ακριβώς για να μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια για την άρση της φτώχειας. Βεβαίω, εκεί αυτό το θέμα αποτελεί θέμα συζήτησης. Τι ακριβώς είναι φτώχεια, πόσα, πόσα ε, κονδύλια μπορούν να διατεθούν, έως ποιο βαθμό θέλουμε να φτάσουμε ε, τους ανθρώπους αυτούς που πλήττονται από τη φτώχεια. Σε κάθε περίπτωση ε, χρειάζεται να αφουγκραστούμε καλύτερα τις ανάγκες των ανθρώπων ε, Ζούμε σε μια εποχή που ακούγονται διάφορες ε, προτάσεις για τη διάθεση κονδυλίων ε, στον ένα τομέα ή στον άλλο τομέα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και χρειάζεται και λογοδοσία και ε, εποπτεία για τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται τα ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε ε, με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ανάγκες ανθρώπων που βρίσκονται, ε, που έχουν πληγεί από αυτήν την ε, ανθρωπιστική κρίση. Θα έχουμε λοιπόν ευρύτατη συνεργασία και με άλλες οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς, ώστε η δράση μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική να τονίσω τέλος ότι υπάρχει και ένα παγκόσμιο σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας. 50% ε, των, της ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίω παρέχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Τέλος, πρέπει να ε, ε σας διαβεβαιώσω ότι παρά τις δυσκολίες εμείς θα συνεχίσουμε στεναρά στο δρόμο που έχουμε χαράξει τον δρόμο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναπτυξιακή βοήθεια. Οι χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν ε, σημαντικά ε, σε αυτόν τον τομέα αν και υπάρχει κίνδυνος τα πράγματα να ανατραπούν. Ε, τα επόμενα χρόνια και υπό το φως του Brexit. Αυτό που χρειαζόμαστε ε, σε κάθε περίπτωση είναι αμεροληψία ε, όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Αναφέρθηκα και στα ζητήματα γραφειοκρατίας είπε ο κύριος Γκέρονς ότι δεν επιτρέπεται να μιλούμε για την αναπτυξιακή βοήθεια παρά μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ δυστυχώς δεν ευθύνομαι για το γεγονός ότι το σύστημα έτσι είναι. Είμαι παρόλα αυτά όμως στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο έργο, οργανωτικό, προκειμένου να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ε, είναι προφανές αυτό. Ε, και παρά την περιπλοκότητά του πρέπει να σας πω ότι το σύστημα που έχουμε θέσει σε εφαρμογή αποφέρει αποτελέσματα. Ε, κυρία Χάουταλα, δικαίως αναφερθήκατε στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία. Όπως γνωρίζετε όλοι, η Συρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια ε, ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της πλήρους ε, ε, πολεμικής σύγκρουσης καθώς συνεχίζονται κάποιες περιφερειακές συγκρούσεις και στην πλήρη κατάπαυση του πυρός που ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί μετά και τη διάσκεψη της Γενέβης όταν και θα δοθεί η δυνατότητα επιστροφής σε πολλούς Σύριους πρόσφυγες στις εστίες τους δεν μπορώ να σας πω πόσο θα κοστίσει, θα μας κοστίσει ε, να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στους 4,8 ε, εκατομμύρια Σύριους που έχουν ε, εκτοπιστεί. Πρέπει να συνυπολογίσετε τα χρήματα που δαπανούν ο Λίβανος και η Τουρκία. Αυτό που επίσης θα έχουμε σε κάθε περίπτωση κατά νου ε, είναι τα ζητήματα και ε, της διαδικασίας της ανικοδόμησης ε, της χώρας, της συμφιλίωσης έπειτα από έναν σημαντικό εθνικό διχασμό που έχει δεχθεί η χώρα αυτή και της επιστροφής βεβαίως των μεταναστών γιατί εφόσον οι μετανάστες αυτοί δεν επιστρέφουν στις αιστείες τους θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Αυτοί ε, είναι και οι άνθρωποι που ε, πολλές φορές ε, περιμένουν οι ίδιοι προσωπικά με τα κλειδιά στο χέρι να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να πάνε ε, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Αυτή είναι και η ανθρώπινη διάσταση ε, της, ε, ε, των θεμάτων αυτών που συζητούμε σήμερα εδώ. Κατανοούμε την σοβαρότητα και την επιτακτικότητα της κατάστασης. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο και γνωρίζω ότι και η ύπατη εκπρόσωπος ε, έχει έλθει σε επαφή και με περιφερειακούς και διεθνείς ε, φορείς και οργανισμούς προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή ε, θα βαίνει βελτιούμενη από εδώ και στο εξή. Δυστυχώς δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς να σας δώσω. Γνωρίζετε όμως ότι η διαδικασία αυτή θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ κοστοβόρα. Ναι, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα και ζητήματα, λέει η Πρόεδρος, ε, και βεβαίως θα πρέπει να δούμε το θέμα της ανοικοδόμησης της ε, ε, Συρίας. και μπορεί όλοι να λένε πρέπει να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα είναι η μόνη. Η Άννη... Α, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσίασή σας. Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις ε, ε, λόγω και της ε, ε, της χώρας σας, ε, της γεωγραφικής, ανάμεσα στην Αφρική και στην Ευρώπη και τις ευθύνες που έχετε επομιστεί εδώ και δεκαετίες ε, για τη διαχείριση της πολιτικής μετανάστευσης. Πράγματα που πολλές βορειοευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν καν κατανοήσει στο σύνολό τους. ακούστηκε από δημοσιογραφικούς κύκλους ότι η Μαλτέζικη Προεδρία έχει διανύμει ε, ένα έγγραφο βάσει του οποίου υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια όσον αφορά την διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα. Ε, ε και στο έγγραφο αυτό ε, ε, επικρίνονται διάφορες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες κατηγορούνται ότι στην ουσία προσελκύουν προς πρόσφυγες και μετανάστες. Εγώ πρέπει να σας πω ότι υποστηρίζω το έργο αυτών των οργανώσεων λόγω και του πολύ σημαντικού αποτελέσματος που έχουν αποφέρει όσον αφορά τη διάσωση ζώων, ανθρώπινων ζώων. Όσον αφορά το πουλς, ε, ε, είχαμε καταφέρει ε, πρόσφατα στο Συμβούλιο ε, να ε, δημιουργηθεί μια κλίδα κατανομής ε, προκειμένου να μην επομίζονται μόνο οι χώρες Νοτιού Ευρώπης με τα προβλήματα που φέρει μαζί της η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Να κλείσω με το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ στην Επιτροπή μας δημιουργεί ε, επισκεφθήκαμε το Emergency Response Coordinator, το κέντρο εκείνο που βοηθά στο συντονισμό της, ε, των φορέων παροχής ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Εκεί λοιπόν μας εξηγήθηκε ότι δεν έχουμε φορητό νοσοκομείο εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν μπορούν να καλύπτονται οι το, το κόστος λειτουργίας παρά μόνο το κόστος μεταφοράς. Μήπως θα μπορούσατε αυτό να το αναλάβετε, να αναλάβετε μια πρωτοβουλία ε, και να βελτιωθεί η κατάσταση. Όσον αφορά το 0,7% το Brexit ε, πρέπει να σας πω ότι ε, το, η Βρετανία ήταν ε, κάποιες από τις ελάχιστες χώρες που ε, νομικά έχει ε, καθορίσει το 0,7% για την ανθρωπιστική βοήθεια και να θέσω και ένα τελευταίο θέμα εμείς είχαμε ζητήσει ως ομάδα αντί για 2% 4% να είναι το ποσοστό που θα κατευθύνεται στην παιδεία για τους πρόσφυγες Αυτά και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην ε, Προεδρία σας. Η Τερέζα Χιμένες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί δυστυχώ δεν μπορούσα να ε, είμαι εδώ τη στιγμή της εκλογής σας. Ήμουν σε άλλες ε, επιτροπές. Να σας συγχαρώ λοιπόν για την εκλογή σας και να συγχαρώ για την αναλυτική του παρουσίαση των ε, ε, Υπουργό της ε, ε, Μάλτας. Να υπενθυμίσω το σημείο 16 των βιώσιμων στόχων, αναπτυξιακών στόχων που αναφέρεται στην ειρήνη και την ανάπτυξη σε χώρες όπως η Νιγηρία ή η Σομαλία, τις οποίες επισκεφθήκαμε στα πλαίσια των χωρών ΑΚΕ. Μόλις γυρίσαμε, εγώ και μερικοί συνάδελφοι άλλοι από τον Αϊρόμπι και είδαμε πώς ζουν το θέμα της τρομοκρατίας και πώς αισθάνεται εγκαταλελειμμένος ο κόσμος εάν δεν υπάρχει ε, σωστή διακυβέρνηση σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και η ανθρωπιστική βοήθεια δύσκολα φτάνει στα σωστά χέρια. η τρομοκρατία τύπου Μπόκο Χαράμ και τα λοιπά υπάρχει ε, και ε, λόγω της διαφθοράς που υπάρχει σε αυτές τις χώρες ε, η επιρροή της είναι ακόμα μεγαλύτερη. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά και πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες αυτές έτσι ώστε ε, να έχουν μια διακυβέρνηση η οποία να ρυθμίσει την ε, φτώχεια και τα, όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία στον κατάλογο, αλλά ιδιαίτερος άξια η συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ ε, και εσάς κυρία Πρόεδρε και τον κύριο Υπουργό. Ε, εκτίμησα πολύ θετικά την συνολική σας αναφορά στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτής της μακροσκελής ε, ε, ερωτήσεις που ήδη υπέβαλαν οι συνάδελφοι και στις οποίες ήδη εκτενώς επίσης απαντήσατε. Ασχολούμαι πάρα πολύ και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην οποία είμαι μέλος, ασχολούμαι λέω πολύ με μετανάστες, πρόσφυγες κλπ. Ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπουμε πάντα από κοινού ε, τις εξελίξεις στη μετανάστευση μαζί με τις εξελίξεις ε, για την ανάπτυξη και μια και είναι επίκαιρα τα στοιχεία αυτά, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς είναι, οι, τι διαστάσεις παίρνουν οι ανθρωπιστικές ε, κρίσεις ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνω υπόψη μου, ας πούμε, τα όσα διαδραματίζονται σε ορισμένα νησιά της Ελλάδας, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Σερβία. Ε, δεν έχουν αρκετά τρόφιμα, αρκετή τροφή, ζουν μέσα στο κρύο σε σκηνές και αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά είναι ότι είδα πάρα πολλούς ανθρώπους χωρίς παπούτσια. Ε, τα συζητήσαμε βέβαια και θα τα ξανασυζητήσουμε και τον Επίτροπο Στυλιανίδη αυτά. Ε, είμαστε πολλοί που ρωτούμε πάντα την Κομισιόν τι μπορεί να κάνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να στραφώ προς το Συμβούλιο. Τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο ε, σε απέναντι σε τέτοιες ανθρωπιστικές κρίσεις. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους λόγω του ψύχους στην προσπάθειά τους να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, ε, κάνουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες. Η Κομισιόν πέρσι κινητοποίησε, ενεργοποίησε μάλλον ένα εργαλείο για τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι αυτό, θα πρέπει, αυτό το εργαλείο θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα το πούμε αυτό στον Επίτροπο Στυλιανίδη αλλά και τα κράτη-μέλη και γι' αυτό στρέφομαι προς εσάς ε, μέσω των εκπροσώπων τους ε, θα πρέπει να είναι περισσότερο παρόντα και κυρίως να βοηθήσουν τις χώρες οι οποίες από μόνες τους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Υπουργέ να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. μου κάνετε ερωτήσεις, ε, ασχολείστε, δίνετε ε, δεδομένα, στοιχεία, όπως έκανε και η τελευταία ομιλήτρια. Ο κύριος Λέτς αναφέρθηκε στην Αφρική. Πολλά έχουμε πει και έχουν υποθεί σχετικά τι θα μπορούσε να σημαίνει η Αφρική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να βοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτής ε, της ε, Υπήρου και μάλιστα γρήγορα. Υπήρξε και ένα ερώτημα σχετικά με πρόταση της Επιτροπής, ε, η οποία θέλει να βοηθήσει, να σταματήσει τους πρόσφυγες να σας πω ότι υπήρξε σήμερα μια κοινή ε, μια κοινή συνέντευξη τύπου των Μογκερίνη και Αβραμόπουλου για το θέμα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν προσπαθούμε να κουκουλώσουμε έτσι με λίγα καλά τα πολλά αρνητικά. Αλλά δεν θέλουμε επίσης να μειώσουμε συνειδητά τα, τους αριθμούς αυτών που ε, προτίθενται να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πάντα σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες των ΕΕ, καθώς επίσης και με την υπηρεσία μετανάστευσης ε, να δούμε τι εφαρμόζεται ε, και αν εφαρμόζεται σωστά η συμφωνία με την Τουρκία και να παρακολουθούμε και την κατάσταση στη Λιβύα. Δεν μπορώ βέβαια να αναλάβω δεσμεύσεις εδώ, πάντως πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ε, η εργασία και τα συζητούμε όλα τα θέματα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ή μια πρωτοβουλία η οποία όμως να μην συμμορφούνται ε, πλήρως ε, με το νομικό ε, πλαίσιο, το υφεστάμενο νομικό πλαίσιο, αλλά και να μην έχει σαν κύριο μέλημα την κάλυψη των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών, που ούτε θέλουμε να πνιγούν στη Μεσόγειο, αλλά ούτε θέλουμε και να γυρίσουν πίσω σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για αυτούς. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πρέπει να δω και την, και την ανταπόκριση των ε, επιτρόπων ε, μετά από την ε, μελέτη αυτή. Τώρα, κοιτάξτε, σχετικά με αυτούς που χάνουν τη ζωή τους στην Μεσόγειο, το ένα είναι να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να μην πνίγονται. Το δεύτερο είναι και σύμφωνα με το σχέδιο Αβραμόπουλου ε, να μπορέσουμε να βρισκόμαστε στα όρια των χωρικών μας υδάτων, γιατί δεν έχουμε ακόμα την ε, νομική δυνατότητα να προχωρήσουμε πιο κοντά στις ακτές της Λιβύης, να μείνουμε ε, εκεί λοιπόν έτσι ώστε ε, να δίνουμε και βάρκες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι και οπωσδήποτε θα πρέπει μετά να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι άλλο είναι να είμαστε γρήγοροι ε, στον διαχωρισμό των ανθρώπων που είναι επιλέξιμοι για ε, υποβολή ε, αίτηση ασύλου και οι υπόλοιποι να επιστρέφονται με γρήγορες διαδικασίες στις χώρες τους. Κοιτάξτε, έχουμε ας πούμε υπογράψει ε, μια συμφωνία με το Μαλί. Ε, αλλά βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μετανάστες από το Μαλί, διότι η κυβέρνηση του Μαλί δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες ε, οι οποίες απορρέουν από την υπογραφή. Δεν μας δεν θέλουμε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιλέξιμος για άσυλο να μην έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα ασύλου. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Ε, τώρα, το θέμα κατανομής Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων οι ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν. Το έχω πει και το ξαναλέω. Όταν συζητήθηκε η αρχή της ε, πραγματικής ουσιαστικής ε, ε, αλληλεγγύης ήταν σαφές ότι πρέπει να μιλάμε για αλληλεγγύη και το επίθετο δεν είναι απλώς κοσμητικό, πρέπει να είναι πραγματικά αποτελεσματική αυτή η αλληλεγγύη. Δυστυχώς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, μία από τις χώρες οι οποίες ε, συμβάλλουν περισσότερο ε, στο, και οικονομικά για τις αντιμετώπιση της μετανάστευσης ενώ υπάρχουν και χώρες ε, οι οποίες όπως η Ιταλία ή η Γαλλία θεωρούν ότι τα χρήματα τα οποία δαπανούν θα πρέπει να συνυπολογίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του ΩΣΑ. Η κυρία Χιμένες αναφέρθηκε στην κυβερνησιμότητα και την ειρήνη. Αναφερθήκατε στην Ιγυρία και στη Δυτική Αφρική γενικά. Μπορώ να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς εδώ ε, ε, μπαίνουμε στο σκέλος της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και συνδέεται και με αυτά τα οποία έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις συμφωνίες, καθώς επίσης και το περιεχόμενο των συμφωνιών με τις χώρες της υποσαχαρίας Αφρικής. Ε, αναφερθήκατε στην ε, ε, Νιγηρία, μα είναι μία μόνο από τις χώρες η οποία, είναι, η οποία μπορεί να αυξήσει τον πληθυσμό της τρομερά τα επόμενα χρόνια. Και έχετε δίκιο ότι το ζήτημα του Μπόκο Χαράμ είναι πολύ σημαντικά και στην Ιγυρία και στη χώρα του Νίγηρα. πραγματικά υποφέρουν οι πληθυσμοί εκεί. Οπωσδήποτε ε, ε, θα θα δώσουμε πολύ μεγάλη ε, συμφωνία στο ΑΓΑΔΙΤΣ, γιατί είναι σημείο περάσματος προς την Λιβύη. Είναι προφανές επίσης ότι εάν κανείς μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει και για ε, αναπτυξιακή βοήθεια και μιλάει και οπωσδήποτε και για τρομοκρατία. Το ένα εξαρτάται από το άλλο και το ένα βασίζεται στο άλλο. Ε, στην Ιταλίδα συνάδελφο, τι να πω, βεβαίω συμφωνώ με αυτά που λέτε και κατανοώ πλήρως ε, την, ε, όχι την έκπληξή σας, αλλά πραγματικά καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε όλες αυτές τις οργανώσεις και να δεχόμαστε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά, τα οποία ε, περπατάνε εξυπόλυτα μέσα στο χιόνι. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά πραγματικά μας συγκινεί τρομερά το να βλέπουμε αυτό το θέαμα. Και τους επόμενους μήνες ε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να υπάρξουν συμφωνίες μεταξύ των χωρών. Τι να σας πω τώρα. Αυτή είναι μία μαύρη κοιλίδα στην συνείδηση της Ευρώπης γιατί ξέρουμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους οι περισσότεροι είναι γυναίκες, παιδιά και νεαροί. Και πρέπει να ε, τους ε, ε, επικουρήσουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους συνδράμουμε αν θέλουμε να ονομαζόμαστε άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι εκτίμησαν όλος ιδιαίτερος ε, τα θέματα που θέσατε ε, οι συνάδελφοί μου. Ε, θα προσπαθήσουμε κατόπιν της συνόδου, της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου να προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους. Πράγματι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεργαστούμε μαζί σας κατά τους ερχόμενους έξι μήνες. Συνάδελφοι, παρακαλώ όσοι αποχωρείτε, αποχωρήστε και οι υπόλοιποι να καθίσετε παρακαλώ, γιατί έχουμε ένα ακόμη θέμα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη συνεδρία των συντονιστών και είναι η έκθεση από την αποστολή μας στην διάσκεψη Habitat 3 ε, που έγινε τον Οκτώβριο από τον κύριο Φολσουρίκα, ε, ο Μπόγκταν, ο Άνταμ και ο Ιγνάθιο συμμετείχαν επίσης ε, και συμμετείχαν και από την Επιτροπή Ρέτζι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σου δώσω το λόγο να το παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες για την ε, σημασία που δίνουν ε, στην ε, ανάπτυξη του οικοσυστήματος στον κόσμο. Η UN Habitat έκανε ε, την, ε, την συνάντησή της τον Οκτώβριο ε, στο Κίτο του Εκουαδόρ. Περίπου 200 αντιπροσωπείες υπήρχαν και αν θυμάστε 40.000 ήταν οι συμμετέχοντες αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προερχόταν από το Εκουαδόρ ε, ο σκοπός ήταν να υπάρξει μια ευρύτερη ατζέντα και ο τρόπος ε, να την ε, εφαρμόσουμε ε, η ανάπτυξη των άστεων είχε ως αποτέλεσμα ε, την απερίμωση ορισμένων περιοχών αλλά δεν κατάφερε να καλέψει ζητήματα όπως τη συμφόρηση, τη ρήμανση, τη ρήπανση, ε, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τον διαχωρισμό και την δημιουργία ανισοτήτων. Κατά τη γνώμη μας η αστικοποίηση δίνει τη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης περιβαλλοντικής προστασίας επίσης ε, και προκλήσεις και ευκαιρίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω προγραμματισμού, σχεδιασμού, ε, ε, οικονομικού μεταξύ άλλων. 40 άτομα υπό την προεδρία της ε, Κορίνα Κρέτου, όπως επίσης και εκπρόσωποι από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις ε, και μέλη της ε, ΕΟΚΕ συμμετείχαν. Η διάσκεψη Habitat 3 προώθησε τις συζητήσεις μεταξύ των παγκοσμίων ηγετών, των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών από όλο τον κόσμο. Η διάσκεψη έληξε με μια ισχυρή έκκληση για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την υιοθέτηση μιας νέας ατζέντα αστικής, η οποία εγκρίθηκε ε, στην ολοκλήρωση της Ολομέλειας 175 παράγραφοι που συμφωνήθηκαν με συνένεση από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Πρόκειται για ένα περιεκτικό ε, έγγραφο ε, συνοπτικό ε, το οποίο σκοπό έχει να ε, καθοδηγήσει τους, τα επόμενα 20 χρόνια αστικής ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και επικεντρώνεται κυρίως σε οικονομικά σε οικονομική ευημερία, κοινωνική ένταξη, ανθεκτική, υγιή πόλη, υγιής πόλη σε όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων, κοινωνίας του πολίτη και και τοπικών ε, κοινωνιών. η, Ευρωπαϊκή, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση της ατζέντα βασίστηκε ε, στη, ε, στο, στο συμπεράσματα του 12 η Μαΐου η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβει η ατζέντα τις δεσμεύσεις που έγιναν ε, το 2013 για την αηφόρο ανάπτυξη, ε, όπως επίσης ε, και στον στόχο... στο στόχο 11 ώστε να είναι ανθεκτικές και βιώσιμες οι πόλεις, όπως και τους ε, συνδεδεμένους στόχους. Επίσης ανέφερε ότι η νέα αστική ατζέντα θα έπρεπε να ακολουθεί μία προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και να λαμβάνει υπόψη ε, κάποια, κάποιες άλλες δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία των Παρισίων ε, και το σχέδιο δράσης αντί Σαμπέμπα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η νέα αστική ατζέντα έχει περιλαμβάνει περιλαμβάνει πάρα πολλούς αξιέπαινους στόχους. Το θέμα είναι πώς θα τους εφαρμόσουμε, γιατί τα μέτρα που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν την νέα ατζέντα, δεν είναι δεσμευτικά για τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χάρτη πορεία ή πρόγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Συνεπώ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι, τα στόχα, ότι οι στόχοι αυτοί θα εφαρμοστούν και θα εκπληρωθούν. Όμως επαφίεται σε εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε κάθε ε, ευκαιρία που έχουμε να επιμείνουμε ότι αυτό το σημαντικό έγγραφο θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Η νέα αστική ε, ατζέντα προβλέπει έναν μηχανισμό εφαρμογής, στο πρόγραμμα εφαρμογής του ΚΙΤΟ. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμογής ε, συμπεριλαμβάνει εθελοντικές ε, δεσμεύσεις από διάφορους εταίρους που σκοπό έχουν να συμμετέχουν και να ενισχύσουν τα αποτέλεσμα της νέας αστικής ατζέντα και τα αποτελέσματα της διάσκεψης Habitat 3. Ε, αναθεώρηση θα γίνεται κάθε, μέσω εκθέσεων θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια την 72η Γενική Συνέλευση το, του ΟΗΕ ε, εντός αυτού του έτους θα υποβληθεί η πρώτη έκθεση ε, η αποστολή μας συμμετείχε σε πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό της διάσκεψης Habitat 3, ε, μεταξύ των οποίων ε, κάποιες είχαν οργανωθεί από τη Regio και την DEFCO. Το, το, το, όπου προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τις δικές μας ιδέες και το δικό μας προφίλ, ε, το, τα, Ηνωμένα, τα Έθνη αγνόησαν την έκκληση από ευρωβουλευτές ε, να ε, πάρουν το λόγο στην συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΟΗΕ. Ίσως θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο στο μέλλον σε κάποιες συνεδριάσεις εδώ που θα έχουμε προσκαλέσει εκπροσώπους του ΟΗΕ πλαίσιο του Habitat 3 ε, συναντήσαμε την Μαριάν Φανστίν ε, και το, την Καμπριέλα Ρίβα Ντενέιρα που είναι η πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Εκουαδόρ Είχαμε μία πάρα πολύ καλή συνομιλία και οι δύο συνεδριάσεις μας έδωσαν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική, οικονομική ε, και κοινωνική κατάσταση στο Εκουαδόρ εν ώψη της ε, των επερχόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που θα λάβουν χώρα στις 19 Φεβρουαρίου του 2017. Ο πρώτος γύρος θα είναι τότε. Η ιδιαίτερη μνήμα έγινε επίσης ε, και στην προσχώρηση του Εκουαδόρ στην εμπορική εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Περού και Κολομβίας ε, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου θα ήθελε επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο ΚΙΤΟ για την υποστήριξή τους στην συμμετοχή και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμες ε, συνεδριάσεις που μας έδωσαν πάρα πολύ καλές ε, πληροφορίες εκ των έσω. Θα ήθελα να ακούσω και από τους άλλους συναδέλφους, αν συμφωνείτε κυρία Πρόεδρε, να μου πούν και εκείνοι αν θέλουν κάτι να πούν. Ο Ιγνάθιο θέλει κάτι να πει. Μπόγκταν, εσύ πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Φραντσουλίτσα. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε σχετικά με τη διάσκεψη του Κίτο και την παραμονή σας εκεί. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα έτσι, επικέντρωσα την προσοχή μου στις ε, συνεδριάσεις ε, οι οποίες αφορούσαν θέματα ε, που μας απασχολούν και εδώ, κυρίως ανάπτυξη και πρόσφυγες επίσης. Ε, ασχολήθηκα και με τις εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή στέγης σε αναπτυσσόμενες χώρες, χώρες. Και τέλος με τις εξελίξεις όσον αφορά τις αστικές ε, περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά ε, σε ε, προστατευόμενες περιοχές, κυρίως δε την άναρχη αύξηση των πόλεων στις άκρες των οποίων ε, δημιουργούνται οι παραγκουπόλεις. Ε, και αστική ε, και ανάπτυξη αστικού ιστού που καμία σχέση δεν έχει με τις αρχές που, έχει ορίσει τα, που έχουν ορίσει τα Ηνωμένα Ελπίζω ότι χάρη στην διάσκεψη θα γίνουν καλύτερα κατανοητές οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοιες παραγκουπόλεις και σε υποβαθμισμένες ε, περιοχές και ότι γενικώ θα υπάρξει βελτίωση της ε, ζωής τους μέσα από βελτίωση των συνθήκων που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές. Ε, επίσης ε, σημαντικό είναι ε, να ασχοληθούμε με ανθρώπους οι οποίοι ζουν κοντά σε εμπόλυμες ζώνες. Ας πούμε να δούμε περιπτώσεις όπως αυτή της Ιορδανίας ε, γιατί η Ορδανία είναι μια χώρα η οποία έχει υποδεχθεί πάρα πολλούς πρόσφυγες από την ε, ε, γειτονική Συρία και επιτρέπει στα παιδιά των Σύρων προσφύγων να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα σχολεία κτλ. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε που μας εκπροσωπήσατε. Ευχαριστώ πολύ ο Ιγνάτσιο πω δύο λόγια ε, αναφερόμενος στην ε, εμπειρία μας ε, στο ΚΙΤΟ χωρίς να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο Σάνσβος Φραντζούλικα και τα οποία προσυπογράφω. Δεν ξέρω εάν όλοι οι συνάδελφοι έχουν ακριβώς την ίδια άποψη με εμένα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμένα δεν με ικανοποίησαν. Ήταν μια χαοτική διάσκεψη ε, διάφορες έτσι, χαοτικές καταστάσεις όπου ε, ε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις για τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί ε, στα αστικά κέντρα. Πολλές συνεδριάσεις ταυτόχρονα, πολλά πράγματα για τα οποία γινόταν συζήτηση ταυτόχρονα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς μια σειρά προτεραιοτήτων. Ήταν δύσκολο να εγγραφεί κανείς και να παρακολουθήσει, δύσκολο να φτάσει μέχρι το τέλος της διάσκεψης έχοντας ας πούμε μια πιο συγκεκριμένη εντύπωση και ιδέα για το περί τίνος πρόκειται. Η... Τέτοιου είδους ε, ε, οργανώσεις από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω αν επιτυγχάνουν το στόχο τους, γιατί αυτή η κατάσταση στην ουσία εκμηδενίζει τις καλές προθέσεις. Ε, δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι συμμετέχοντε είχαν άλλη ε, εντύπωση και αποκόμισαν διαφορετικέ εντυπωσει. Εγώ σας λέω τα δικά μου. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γκαμπριέλ Ονάκα. Θέλετε να λάβετε τον ε, λόγο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνδιάσκεψη Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη τη αντιπροσωπεία τη ε, ε, Επιτροπή ε, Ανάπτυξη που συμμετείχαν παρά το χαοτικό πρόγραμμα και το πολύ ευεβαρημένο πρόγραμμα και όσον αφορά το τμήμα της DigiRegio. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή για τα συμπεράσματα ε, σχετικά με την εργασία που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε γενικές γραμμές ε, η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη όσον αφορά το πρόγραμμα, όσον αφορά το περιεχόμενο του νέου προγράμματος και του νέου θεματολογίου. Για το γεγονός ότι ε, μεγάλος αριθμός των συμπερασμάτων του Συμβουλίου στην ουσία επιβεβαιώνουν τις ε, αρχές ε, αυτές. Βεβαίως ε, παραμένουν ακόμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν, κυρίως όσον αφορά ακριβώς την υλοποίηση των προγραμμάτων και για την Κομισιόν αλλά και για τις, τα υπόλοιπα όργανα, τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κεντρικές κυβερνήσεις, τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις όσον αφορά την υλοποίηση. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν ήδη άρχισε να εργάζεται επί τριών εθελοντικών δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί και που παρουσιάστηκαν στο Κίτο από, το, από την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπη κ. Κορίνα Κρέτσου. Να πω ότι όσον αφορά ε, στην ε, συμβολή ε, του νέου θεματολογίου μέσω της ε, υλοποίησης ε, και της εφαρμογής του αστικού θεματολογίου. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Βάσει αυτού λοιπόν ξεκινήσαμε 8 εταιρικέ σχέσεις πέρσι και φέτος, 8 από τις 12 που περιλαμβάνει το αστικό θεματολόγιο. Σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις έχουμε εκπροσώπους πόλεων, αστικών αρχών, ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επίσης εκπροσώπους της Κομισιόν. Αυτές οι εταιρικέ ε, σχέσεις ε, εντός τριών ετών θα υλοποιήσουν σχέδια δράσης τα οποία στόχο έχουν την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, την βελτίωση της χρηματοδότησης καθώς επίσης και την καλύτερη γνώση των βελτίστων πρακτικών και ανταλλαγών των ιδίων μεταξύ των αρχών. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, multi-level governance, σε επίπεδο λοιπόν εθνικής, τοπικής, περιφερειακής διακυβέρνησης αλλά και ενωσιακής εμείς στα πλαίσια αυτών των ε, εταιρικών σχέσεων. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε και να διασφαλίσουμε μάλλον ότι οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ε, προκλήσεις σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες περιλαμβάνονται ε, στην νέα, στο νέο αστικό θεματολόγιο, αλλά και κάποιους στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στο, στην Ατζέντα 2030, διασφαλίζοντας την συνεκτικότητα και τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και ε, διεθνές πλαίσιο. Τα πρώτα σχέδια δράσης ε, θα παρουσιαστούν φέτος το καλοκαίρι. Τέσσερα σχέδια δράσης λοιπόν θα παρουσιαστούν ε, μετά περί τα μέσα της επόμενης ε, χρονιάς θα έχουμε και άλλα τέσσερα ε, σχέδια δράσης και τέλος περί τα τέλη του 2018 θα έχουμε τα τέσσερα τελευταία σχέδια δράσης που θα καλύψουν εν τέλει και τα 12 θέματα, τους 12 τομείς του θεματολογίου, του αστικού θεματολογίου και που θα καλύψουν ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις της Ατζέντα 2030. Όσον αφορά τις άλλες δεσμεύσεις του Κομισιόν, πρόκειται για, αναφέρομαι εδώ, σε μια πιο τεχνικής και επιστημονικής φύσεως δέσμευση, ε, αφορά την συνολική και εναρμονισμένη, συγγνώμη, τον συνολικό και εναρμονισμένο ορισμό ε, της... Ε, ε, της μετανάστευσης και εδώ έχουμε από κοινού δουλέψει με τον Όσα και την Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε ε, να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης με ρόλους ε, και επιδιώξεις ρητά ε, σταθμισμένες. Ε, το 2017 ε, θα έρθουμε σε επαφή με τις στατιστικές υπηρεσίες ε, κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χώρες όσα, έτσι ώστε να δούμε ποιες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν βάσει του συνολικού πληθυσμού. Το 2017 θα ξεκινήσουμε πιλωτικά προγράμματα με τις ε, στατιστικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας υφιστάμενα ε, στοιχεία για να δούμε το συσχετισμό των πληθυσμών και τέλος ε, την επόμενη χρονιά θα τροποποιήσουμε τον ορισμό της αστικοποίησης ε, υπό το φως των νέων στοιχείων. Και το 2019-2020 ε, θα είμαστε πλέον σε θέση να ε, προτείνουμε στη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών ένα ορισμό που θα είναι αποδεκτός από όλους. Στο τρίτο στοιχείο βρισκόμαστε ήδη ε, σε διοικητική προπαρασκευή για την συνένωση και από κοινού αντιμετώπιση των ισοτικών περιοχών. Ναι, συγγνώμη που σας βιάσα λίγο, αλλά έχουμε συνεδρίαση συντονιστών. Θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω ε, ε, όλους όσους συμμετείχαν στην αποστολή αυτή και που έλαβαν το λόγο. Ε, πρέπει βεβαίως να δοθεί συνέχεια στο θέμα αυτό και να το ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και με αυτό κηρύσω τη λήξη της τακτικής μας συνεδρίας. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ε, η συνέδριση των συντονιστών θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Αφού αποχωρήσουμε.